Περνάμε στην κοινή συνεδρία των δύο επιτροπών μας. Η συνεδρία ξεκινάει τώρα και θα συνεχιστεί αύριο στις 11. Πρώτα απ' όλα έγκριση της ημερησίας διάταξης. Εντάξει βλέπω. Δεν έχουμε ανακοινώσεις ε, του Προέδρου. Πάμε κατευθείαν στο πρώτο σημείο. Η δημιουργία Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου Εισηγητή Πέντρο Σίλβια Περέιρα και Βλαντιμίρ Μπάκαν. Να δώσω τώρα τον λόγο στον συνάδελφο από την Επιτροπή Προπολογισμού που θα προεδρεύσει. Ευχαριστώ. Αναλάβω εγώ λοιπόν την διεύθυνση της ε, συζήτησης. Έχουμε μέχρι τις 7 η ώρα. 45 λεπτά δηλαδή. Να ξεκινήσουμε έτσι κάπως γρήγορα. Τον λόγο έχουν οι δύο εισηγητές. Ε, πρώτος ο Πέντρο Σίλβα Περέιρα. Είναι πρώτος ο δικό μου κατάλογο. Έχεις τον λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Να ευχαριστήσω τον συνσηγητή μου πρώτα απ' όλα τον κύριο Μάνκα για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε στην προετοιμασία αυτού του σχεδίου έκθεσης για το λεγόμενο Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο. Η ιδέα λοιπόν δημιουργίας αυτού του ταμείου δεν είναι καινούρια, έχει συζητηθεί εντόνως τα τελευταία χρόνια στο πλαίσιο της ε, μεταρρύθμισης της οικονομικής και νομισματικής μας ένωσης η πρόσφατη πρόταση της Κομισιόν ε, το Μεκέμβριο του 2017 ε, είναι νομίζουμε καλοδεχόμενη ως μια σημαντική συνεισφορά στην συζήτηση και πρέπει να αντλήσουμε τα διδάγματα της οικονομικής ε, κρίσης να ενισχύσουμε την Ευρωζώνη χρησιμοποιώντας ε, και δημιουργώντας κάποια στιβαρά εργαλεία για να στηρίξουν τα κράτη-μέλη που έχουν ανάγκη για να διασφαλιστεί η σταθερότητα των οικονομιών μας στην περίπτωση μελλοντικών ασύμετρων και συμμετρικών καρδασμών. Βεβαίως και αυτό δηλώνεται καθαρά στο σχέδιο της έκθεσής μας η δημιουργία του μέσου αυτού και μελλοντικά του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας ε, έχουν δημιουργήσει ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση ενός μηχανισμού διαχείρισης κρίσεων και έχουν δώσει οικονομική βοήθεια σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες. Τώρα όμως ήρθε η στιγμή να συζητήσουμε τη μεταρρύθμιση του μηχανισμού σταθερότητα και θεωρούμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να συνεισφέρει σε αυτήν την συζήτηση. Το σχέδιο έκθεσης το οποίο παρουσιάζουμε σήμερα είναι φιλόδοξο αλλά και ρεαλιστικό. Λαμβάνει υπόψη το τρέχον πολιτικό τοπίο έχοντας κατά νου και το μακροπρόθεσμο όραμά μας για το μέλλον. Γι' αυτό η πρότασή μας βασίζεται σε μια απτή προσέγγιση, σε μια απτή πρόοδο, πρόθεσμα, αλλά και στο να αποσαφηνίσουμε τις προτεραιότητες του Κοινοβουλίου μέσω μακροπρόθεσμα. Θα ήθελα να επισημάνω ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να επαναλάβει την ανάγκη να ενταχθεί το μελλοντικό αυτό όργανο στο κοινοτικό δίκαιο, όπως ήδη έχει πει πολλές φορές το Κοινοβούλιο. Ταυτόχρονα και για να διασφαλίσουμε ότι οι νομισματικές λειτουργίες θα είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της Κεντρικής Τράπεζας, το σχέδιο έκθεσης προτείνει μια αλλαγή ονόματος του θεσμικού οργάνου και αντί για Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο προτείνουμε, να το πούμε, Ευρωπαϊκό Ταμείο Σταθερότητας. Είναι έτσι πιο σωστή η ονομασία δεν δημιουργούνται παρεξηγήσεις όσον αφορά την καθανομία αρμοδιοτήτων, δηλαδή η νομισματική πολιτική παραμένει αρμοδιότητα της ΕΚΤ. Δεύτερον, ζητάμε την δημιουργία μια καβάτζα στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Διάσωσης ε, εξυγίανσης, με συγχωρείτε καθώς ε, βεβαίως και την ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασφάλισης ε, Καταθέσεων ε, και θεωρούμε ακριβώς ότι η δημιουργία του ενιαίου Ταμείου Εξυγένσης θα πρέπει να προχωρήσει στο να γίνει αυτό επιχειρησιακό το συντομότερο δυνατόν. Τέλος, για να μην υπάρχει ένας φορέας ο οποίος θα σώζει μόνο τράπεζες, θεωρούμε ότι το βασικό καθήκον αυτού του θεσμικού οργάνου θα πρέπει να είναι η στήριξη στα κράτη-μέλη στην περίπτωση σοβαρών οικονομικών κρατασμών. Επίσης, ξεκαθαρίζουμε ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει άλλη επικάλυψη μεταξύ των αρμοδιοτήτων αυτού του θεσμικού οργάνου και της δημοσιονομικής εποπτείας που κάνει ίδια η Κομισιόν. Και τέλος κύριε Πρόεδρε, θεωρούμε ότι υπάρχει βραχυπρόθεσμα περιθώριο να εισαχθούν κάποιες βελτιώσεις όσον αφορά την σχέση μεταξύ του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας και του Κοινοβουλίου αυτού όσον αφορά ειδικά το θέμα της δημοκρατικής νομοποίησης και λογοδοσίας. Ακριβώς για να υπάρξει υπεραιτέρω κα, κατεπίγουσα εμβάθυνση της οικονομικής διακυβέρνησης της Ευρωζώνης. Αυτές είναι οι προτάσεις μας και τώρα αναμένουμε την άποψη των συναδέλφων για να συνεισφέρει θετικά το Κοινοβούλιο σε μια πολύ σημαντική συζήτηση που αφορά τη μεταρρύθμιση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Τον λόγο έχει ο συνάδελφος Μάνκα, ο συνεισηγητής. Ευχαριστώ, pekne, pán predseda. Chcem sa poďakovať ε, Pedrovi Θέλω να ευχαριστήσω τον συνάδελφό μου, τον Πέδρο Περέιρα. Είχαμε πολύ καλή συνεργασία, έκανε πάρα πολύ καλή σύνοψη, οπότε θα είμαι και εγώ σύντομα στη χώρα μου τη Σλοβακία. Λόγω και του Συμφώνου Σταθερότητας, ε, την έπεσε η κυβέρνηση και Είχαμε ψηφίσει για το αν θα πρέπει να στηρίξουμε το ευρώ, την Ελλάδα κτλ. Και αν δεν είχε δημιουργηθεί αυτός ο μηχανισμός και σε διακυβερνητικό επίπεδο θα είχαμε πολύ βαθιά προβλήματα. Αυτό ήταν ε, η κατάληξη. Δηλαδή τελικά συνειδητοποιήσαμε ότι είναι σημαντικό να υπάρχει μια ισχυρή ευρωζώνη για όλα τα μέλη ε, της Ένωσης και όχι μόνο για όσους είναι στην ευρωζώνη. Αυτό ήταν ένα μεγάλο μάθημα, ένα καλό μάθημα και για μας. Δεν μπορεί κανείς να δίνει μόνος του τις μάχες γιατί αυτό μπορεί να έχει κακό αποτέλεσμα και για αυτόν που αγωνίζεται αλλά και για όλους τους άλλους. Άσε που υποστηρίζουν, ε, έτσι, ε, υποστηρίζονται οι λαϊκιστές. Εμείς θέλουμε αλληλεγγύη και στενή συνεργασία στην Ευρώπη. Τι δημιουργούμε εδώ τώρα. Σε ό,τι αφορά τις δημοσιονομικές πτυχές, Θέλω να πω ότι στο μηχανισμό σταθερότητας περιλαμβάνονται ε, τα κράτη-μέλη τη Ευρωζώνη με το νέο, ακόμα και με το νέο ταμείο που θέλουμε να δημιουργήσουμε, θα καλύπτονται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης οι ζημίες. Δηλαδή, αυτό που πρέπει να δούμε είναι αν θα κάνουμε θα συνδέσουμε τον προπολογισμό αυτό το νέο με την έγκριση του προπολογισμού εν γέννη. Το ελεγκτικό συνέδριο μιλάει για κάποιες διακυβερνητικές λύσεις που μόνο έκτακτες όμως θα πρέπει να είναι. Καλύτερα να εφαρμοστεί η κοινοτική μέθοδος. Άρα στηρίζει τα μέτρα που προτείνουμε και το ελεγκτικό συνέδριο. Και ο τρέχον μηχανισμό, αλλά και ο νέο δεν πρέπει να χρηματοδοτούνται από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό. Για μας προϋπόθεση είναι να μην συμβαίνει κάτι τέτοιο. Θα πρέπει στην ιδρυτική πράξη, στο καταστατικό, να περιλαμβάνονται όλες οι σχετικές διατάξεις Αυτά νομίζω αρκούν ως εισαγωγή, αλλά θα ήθελα να ακούσω και τους συναδέλφους μου τι έχουν να πούν. Ähm, ευχαριστώ. ευχαριστώ. Να ακούσουμε και τους σκιώδεις εισηγητές. Για το ΕΛΚ, ο συνάλφος Φαντεν Κέντελάρε και μετά ακολουθεί και ο άλλος ε, συνάδελφος. Σας παρακαλώ δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα κάνω ό,τι μπορώ ε, για να σας ε, κάνω μια παρέμβαση αρκετά σύντομα. Ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή. Πράγματι θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα πραγματικό Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο για να αποθαρρύνουμε και τους κερδοσκόπους. Είναι σημαντικό τώρα ω Ευρωκοινοβούλιο να αναμειχθούμε σε αυτή τη συζήτηση και μάλιστα γρήγορα. Υπάρχουν μία σειρά ζητήματα που πρέπει να τονίσουμε περαιτέρω. Θα σταθώ σε πέντε. Πρώτον, για το ΕΛΚ είναι πολύ σημαντικό το Ταμείο αυτό να ε, έχει και διατάξεις πρόληψης κρίσεων και διαχείρισης βέβαια. Πρέπει να δίνει στήριξη για απαραίτητε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στα κράτη-μέλη που θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στην ε, αγορά. Μετά, είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι όταν προβλέπει η ε, οικονομική στήριξη του Ταμείου θα πρέπει να συνδέεται πάντα με αυστηρέ ε, προϋποθέσεις πολιτική. Αυτό ακόμα δεν κατονομάζεται και είναι σημαντικό. Μετά, το Σύμφωνο Σταθερότητα και Ανάπτυξη ε, και η αναφορά του είναι κάτι πολύ σημαντικό για να φτιάξουν από μόνο του τα κράτη-μέλη αναχώματα απέναντι σε τέτοιου κρατασμού. Στην ατολική σκέψη, σκέψη ε, υπάρχει μια αναφορά στην ε, ευθύνη των κρατών μελών, θέλαμε να βοηθηθεί περαιτέρω. Θέλουμε να αυξήσουμε την ε, διαφάνεια για τη λογοδοσία. Είναι σημαντικό να υπάρχει αυτό και ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι πολύ θετικό που το σχέδιο έκθεσης ήδη το αναφέρει. Όμως θα πρέπει να ακούγεται και η φωνή των Εθνικών Κοινοβουλίων σε αυτό το σημείο. Θα θέλαμε να λάβετε αυτό το στοιχείο υπόψη. Το Ταμείο λοιπόν δεν θα πρέπει ε, να περιορίζει με οποιονδήποτε τρόπο τα δικαιώματα ε, και τη λογοδοσία ε, των εθνικών και τον δημοκρατικό έλεγχο μάλλον των εθνικών κοινοβουλίων. Τέλος, είναι σημαντικό ο διοικητή του Ταμείου να επιλέγεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο και να λογοδοτεί σε αυτό. Τέλος, κάποια στοιχεία που πρέπει να διευκρινιστούν, όπως ο προσδιορισμός των αρμοδιοτήτων, το ύψο του Ταμείου. Ποιο θα το καλύψει το πιο σημαντικό. Υπάρχουν τέτοιου είδου ζητήματα που μα ενδιαφέρουν και σίγουρα θα τα συζητήσουμε στο μέλλον. Ο σκιώδης εισηγητής ε, από τους Δημοκράτες, ο κύριος Μούρες, ανοιχτό. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα να συγχαρώ τους δύο συνεισηγητές για αυτή την έκθεση που νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα ε, ισορροπημένη και λαμβάνει υπόψη τις ε, απόψεις που υπάρχουν για αυτό το πολύ σημαντικό θέμα. Κάποιες σκέψεις από πλευράς μου. Πρώτον, είναι πολύ σημαντικό το Ταμείο αυτό να έχει τα απαραίτητα πυρομαχικά. Γιατί όλα είναι θέμα αξιοπιστίας. Γι' αυτό και θα πρέπει να αποσαφινιστεί το θέμα της χρηματοδότησης με πολύ πιστικό τρόπο και προς τους συμμετέχοντες στην αγορά. Δεύτερον, πρέπει να είναι σαφές ότι θα είναι ένα μέσο έκτακτη ανάγκης. Για να είμαστε σε θέση λοιπόν να αντιμετωπίζουμε και να χειριζόμαστε τέτοιες ε, κατεπίγουσες περιστάσεις επίπεδο EMF, Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου, θα πρέπει να επενδύσουμε και στην πρόληψη κρίσεων. Να ενθαρρύνουμε τα κράτη να έχουν ισοσκελισμένους ε, προπολογισμού και το καθεξής. Γιατί θα μπορούσε κανείς να πει ότι δημιουργήθηκε, χτίστηκε ένα νέο νοσοκομείο στη γειτονιά μου. Δεν σημαίνει ότι τώρα ε, εγώ πρέπει να αλλάξω τις συνήθειές μου γιατί δεν με νοιάζει υπάρχει νοσοκομείο. Όχι, πρέπει να έχω ισορροπημένη διατροφή, να πηγαίνω γυμναστήριο, να ασκούμε, απομένως διαφορετικέ μεταρρυθμίσεις εν γέρος, για να μην αρρωστήσω. Παρότι υπάρχει καλό νοσοκομείο και πάλι δεν θέλω να αρρωστήσω. Κάπως έτσι είναι και με το ταμείο αποτελεσματικότητα, διαφάνεια και ε, λογοδοσία, ζητήματα ευθύνης και του Κοινοβουλίου, πρέπει να προσδιορίσουμε περαιτέρω τον ρόλο των Εθνικών Κοινοβουλίων. Λαμβάνοντας υπόψη και τους συνταγματικούς περιορισμούς ορισμένων κρατών μελών. Και να εξετάσουμε και τη συμμετοχή χωρών εκτός Ευρωζώνης θα πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε επί της ενότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να στείλουμε το μήνυμα σε χώρες εκτός Ευρωζώνης ότι δεν μπορούν να συμμετάσχουν ε, σε αυτή τη διαδικασία. Αυτή η άγουσα θα αποθάρρυνε περαιτέρω κρατημέλη από το να ενταχθούν στο μέλλον. Γι' αυτό πρέπει να ε, βρούμε και κάποια λύση για τις χώρες εκτός Ευρωζώνης. Και προσβλέπουμε συνεργασία με τους δύο συνεισηγητές στο πλαίσιο της Επιτροπής μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για το ECR, τώρα συνάδελφος Κόλμελ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αναγνωρίζω ότι εργάστηκαν σκληρά οι δύο συνεισηγητές, αλλά θα μπω τώρα κατευθείαν στην ουσία. Ένα ευρωπαϊκό νομισματικό ταμείο είναι άχρηστο. Γιατί συνεχώς λέμε εδώ πέρα και μου λέτε εμένα ότι είναι επιτυχημένο το ευρώ. Κάθε φορά που λέω κάτι μου λέτε είναι επιτυχημένο το ευρώ. Πώς χρειαζόμαστε κάτι τέτοιο στο δέκατο έτος των πολιτικών διάσωσης του ευρώ. Δεν μπορώ δηλαδή με κάθε καλή βούληση να αναγνωρίσω ποιο είναι το νόημα σε όλα αυτά. Δηλαδή, αν είναι το θέμα η σταθεροποίηση του ευρώ, τα πράγματα είναι απλά φροντίστε να τηρούνται τα κριτήρια του Μάστριχτ. Αυτό είναι σταθεροποίηση. Αλλά εάν ξεχνάμε ότι υπάρχουν τεράστιοι κίνδυνοι, αν δείτε μόνο τους αριθμούς του Target 2, που αυτή τη στιγμή είναι εις βάρος της Γερμανίας ε, ε, σχεδόν ένα τρισεκατομμύριο ευρώ, χωρίς καμία κάλυψη αν δείτε ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εδώ και χρόνια έχει μια πολιτική μηδενικών επιτοκίων, αγοράζει κρατικά ομόλογα, δεν ξημεύσαν σε τίποτα όλα αυτά. Γιατί, γιατί το ευρώ έχει μια εσωτερική αντίφαση. Δεν ταιριάζει δυστυχώς σε όλες τις χώρες που είναι μέλη της Ευρωζώνης. Και εδώ πέρα λέτε ότι με λίγα δισεκατομμύρια ευρώ θα λύσετε το πρόβλημα. Ε, εδώ πρέπει να ομολογήσω ότι πραγματικά ξεπερνάτε τα όρια της αντίληψής μου. Ευχαριστώ. Και φτάσαμε στους φιλελεύθερους. Έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Άκουσα ένα κομμάτι των όσων είπε ο προλαλής σας. Μίλησε για ένα τρισεκατομμύριο στο Target 2 εγώ δεν τα βλέπω τόσο τραγικά τα πράγματα. Ξέρω πως δεν είναι βέλτιστος νομισματικός χώρος η Ευρωζώνη, δεν είναι τίποτα το καινούριο αυτό. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι η προσέγγιση να γίνει ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας σε ένα Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο επί της αρχής είναι σωστή. Εντάξει, πιθανώ. Ε, θα χρειάζεται να έχει το ίδιο όνομα και στο μέλλον γιατί έτσι δεν θα χρειάζεται να κάνει όλες ε, τις αλλαγές για να έχει μια νέα διεθνή αναγνώριση. Προσωπικά λυπούμε για το ότι παρά τις υποσχέσεις ε, το νέο αυτό ταμείο ή μηχανισμό, όπως και να έχει θα παραμείνει διακυβερνητικό. Και μας είχαν υποσχεθεί το αντίθετο όταν ιδρύθηκε. Και πρέπει να πω ότι είχα βασιστεί σε αυτήν την υπόσχεση και τώρα είμαι απογοητευμένο. Θα ήταν νομίζω ένα καλό μήνυμα να δείξουμε ότι το ταμείο αυτό ε, είναι υπεύθυνο σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο, απέναντι δηλαδή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι δυνατότητες βέτο που προκύπτουν από το συνταγματικό δικαίωμα για τα εθνικά κοινοβούλια θα περιέρχονταν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μπορούν να συνεπάρξουν και τα δύο. Σημαντικό είναι να είναι ανεξάρτητο, όπως και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ανεξάρτητο από οποιαδήποτε εθνική επιρροή να κάνει τις αναλύσεις του και να καθορίζει τα προγράμματα μεταρρύθμισης ε, και διάσωσης. Και βεβαίως ε, θα πρέπει, αν θέλει να επιτελέσει την ε, λειτουργία του, να δράσουμε σύμφωνα με το σύνθημα βοήθεια ναι, αλλά μόνο εάν υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα. Αλληλεγγύη ναι, αλλά μόνο με αντάλλαγμα τις αλλαγές. Και βεβαίως αν υπάρξει κάποια παραβία θα πρέπει να έχει και την δυνατότητα κυρώσεων. Και δεν θα πρέπει να περιμένει να έχει την άδεια της Κομισιόν γιατί μέχρι στιγμής έχουμε δει ότι η Κομισιόν δυσκολεύεται να επιβάλλει κάποιες κυρώσεις τις οποίες ε, τις επιτρέπεται οι οποίες τις επιτρέπονται και δεν είναι οπωσδήποτε δυνατόν να πηγαίνουν τα λεφτά των φορολογουμένων για διασώσεις χωρίς καμία διασφάλιση θα πρέπει να ισχύσει η ρήτρα περί μη διάσωσης. Συντομεύεται, λέει ο πρόεδρος. Οπότε αν μια χώρα έχει δυσκολίες θα πρέπει πρώτα απ' όλα να διασφαλιστεί η ε, συμμετοχή των πιστωτών πριν ε, δοθούν χρήματα των φορολογούμενων. Και βέβαια αποφασιστική σημασία είναι η επενδυτική κατηγορία των εθνικών ομολόγων να μην είναι τόσο προνομιούχα ε, στο παρελθόν και έτσι οι τράπεζες θα είναι πολύ πιο προσεκτικές για το αν θα δεχτούν τέτοιου τίτλους. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι και τα κράτη θα αναγκαστούν να είναι πιο φερέγγια γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουν να αντλήσουν χρηματοδότηση από τις αγορές. Είχατε ήδη την ευκαιρία Νομίζω με ακούσατε που είπα δύο λεπτά ο καθένας ε, και έδειξα πολύ μεγάλη υπομονή με τους φιλελεύθερους συναδέλφους. Σας ευχαριστώ. Μάλιστα το εκμεταλλευτήκα τόσο πολύ ώστε δεν βλέπω κάποιον άλλον ε, από άλλη ομάδα οπότε ε, ακούσουμε τώρα τους συναδέλφους τους υπόλοιπους που ζήτησαν τον λόγο δηλαδή την κυρία Μπερέσου ουσιαστικά. Ευχαριστώ. Το βλέπουμε με την ανταλλαγή επιχειρημάτων που προηγήθηκε. Όπως συμβαίνει, μπαίνουμε σε μια συζήτηση χαρακομμάτων. Αντί να αναζητούμε λύσεις, ο καθένας ταμπουρώνεται πίσω από τα επιχειρήματά του, που είναι και άκρος ιδεολογικού χαρακτήρα στη τελική ανάλυση. Και δεν νομίζω ότι λαμβάνουν υπόψη τα διδάγματα που έπρεπε να είχαμε αντλήσει από την κρίση που μας ανάγκασε να υλοποιήσουμε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και παραγνωρίζουν, αγνοούν την εμπειρία που αποκτήσαμε με την λειτουργία αυτού του μηχανισμού. Θέλω να υπενθυμίσω απλά ότι η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ήταν ανέκαθεν ότι ο μηχανισμός αυτός, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας, πρέπει να ενταχθεί στο κοινοτικό πλαίσιο. Με πολλά ψηφίσματα το έχουμε υποστηρίξει. Άρα τώρα που τίθεται το θέμα γυρίζουμε πίσω για την αλλαγή του ονόματος. Είπε ο πρόεδρος Ντράγκη πριν, ο διοικητής Κεντρικής Τράπεζας, ότι για το δικό του το θεσμικό όργανο είναι σημαντικό να μην υπάρχει σύγχυση σε ό,τι αφορά το ποιος ασκεί τις νομισματικές εξουσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είπε ότι συμφωνεί με το ονομασία που προτείνουν οι συνεισηγητές. Αυτό είναι σημαντικό. Τώρα, πώ μπορεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συμμετέχει στη διαδικασία. Εγώ είμαι υπέρ μια θεσμική αρχιτεκτονική που δεν θα είναι και υπερβολικά πολύπλοκη. Έχουμε το μονοπόλιο τη πρωτοβουλία ε, που το ασκεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, παρακολουθεί τη δημοσιονομική πολιτική των κρατών μελών. Αυτή είναι η βάση. Από εκεί και πέρα. Περιμένοντας να μπει στην κοινοτική μέθοδο το, ευρωπαϊκό Μηχανισμό σταθερότητα. να βελτιώσουμε το πλαίσιο διαλόγου, αυτό δηλαδή μεταξύ Κοινοβουλίου και ESM δεν μας δημιουργεί κανένα πρόβλημα. Υπάρχει όμως το ζήτημα της νομιμοποίησης του οργανισμού. Είναι μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία αυτονομίας του οργανισμού, ενώ η προσέγγιση ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί. Τώρα, Ποιε είναι οι δυνατότητε, ποιο είναι το δυναμικό του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας. Ξέρουμε ότι θα ασκεί ε, τη λειτουργία του σε σχέση με το Ταμείο Εξυγείωσης, αλλά θα είναι και ένα backstop ε, για άλλες ε, συμπληρωματικές λειτουργίες που θα τις χρειαστεί ο ναι. Και αν μου επιτρέπετε μια τελευταία λέξη για την κατάσταση των χωρών που δεν ανήκουν στην Ευρωζώνη. Ξέρουμε πολύ καλά ότι το ευρώ δεν θέλουμε να είναι μια λέσχη κλειστή, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να αναλάβουμε όλε τι ευθύνε μας. Οι χώρε που δεν ανήκουν στην Ευρωζώνη θα πρέπει κατά την άποψή μου να αποφεληθούν του Brexit για να πούν ξεκάθαρα πότε και πώς θέλουν να μπουν στην Ευρωζώνη. Ποτέ δεν τέθη αυτό το ερώτημα. Αλλά βαραίνει ε, τις συζητήσεις μας. Εμείς που είμαστε στην Ευρωζώνη και άλλοι που δεν είναι στην Ευρωζώνη, νομίζω ότι μετά τον Brexit πρέπει να είμαστε στην ίδια νομισματική ένωση, στην ίδια νομισματική ζώνη. Σίγουρα υπάρχουν δυσκολίες προσχώρησης, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να επωφεληθούμε του προευλογισμού και του κοινού νομίσματος όλοι. Από την Κομισιόν είστε ευπρόσδεκτοι, λέει ο Πρόεδρος, θέλετε κάποιος από εσάς να πάρει το λόγο. Ναι, ευχαριστώ. Θα τα πω αγγλικά. Ευχαριστώ πολύ. Όσο Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σας ευχαριστούμε για τη στήριξη της πρότασής μας, την οποία εκφράστηκε εδώ και στο σχέδιο έκθεσης. Όπως αναφέρεται και στην πρότασή μας, είμαστε βαθιά πεπισμένοι ότι ε, το Ταμείο έχει ε, αναλάβει σημαντικό ρόλο στο ευρύτερο πλαίσιο διαχείρισης κρίσεων στην Ευρωζώνη. Γι' αυτό και θεωρήσαμε ότι είναι κατάλληλη χρονική στιγμή ε, να ενσωματώσουμε αυτό το σημαντικό διοργανικό φορέα και στο κοινοτικό πλαίσιο. Γι' αυτό και υποβάλλουμε αυτή την πρόταση. Σημειώνουμε όμως ε, και τον πιθανό στόχο να μην αφήσουμε εκτός αυτή την ιδέα, να έχουμε μία ενδιάμεση προσέγγιση οι προτάσεις λοιπόν να γίνονται για ένα ενδιάμεσο καθεστώς μέχρι να εξασφαλίσουμε επαρκή στήριξη ε, για την ε, μεταφορά στο, ευρωπαϊκό πλαίσιο. Για τα μέτρα που προτάθηκαν, να επιστήσουν την προσοχή της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου σε ένα έγγραφο που δημοσιεύτηκε πρόσφατα από τον ESM και την Εκομισιόν με κοινή τους θέσεις, θέση για πιθανούς τρόπους ενίσχυσης του ρόλου και της προβολής του ESM έτσι Το έγγραφο αυτό μπορείτε να το βρείτε ε, στον ιστότοπο της Κομισιόν και του ESM. Εδώ αναφέρουμε και τη στήριξή μας για την αύξηση της διαφάνειας και λογοδοσίας του ESM και υπό τη μορφή του διοργανικού θεσμικού οργάνου και αυτό συνάδει πλήρως με τον στόχο που εξυπηρετούμε με την έκδοση της υποβολή της πρότασής μας και αυτό ανακλάται και ε, στην έκθεση εδώ, γι' αυτό και στηρίζουμε πλήρως ε, την πρόταση αυτή, να βρούμε τρόπους αύξησης Τη λογοδοσία και της διαφάνεια για τον ESM, ε ακόμα και αν προς το παρόν παραμένει ε, διοργανικό θεσμικό όργανο, μέχρι να φτάσουμε στο σημείο να ε, τεθεί σε πλήρες κανονιστικό πλαίσιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Εξαντλήθηκε ο κατάλογος των ομιλητών. Να δώσω τον λόγο στου δύο συγγητές, αν το επιθυμούν. Κύριε Μάνκα. Σίλβα Περέιρα τότε. Ευχαριστώ πολύ. Αρχικά να σας ευχαριστήσω για τα σχόλιά σας. Με τα χαράς βλέπω ότι ε, αναγνωρίζατε ότι πρόκειται για ένα ισορροπημένο σχέδιο έκθεσης και καλή βάση συνέχιση των εργασιών. Πρόθεσή μας ήταν να συμβάλλουμε θετικά στη συζήτηση για την μεταρρύθμιση του ESM. Γι' αυτό και προτείναμε αυτή την ε, προσέγγιση των δύο βημάτων. Μακροπρόθεσμα θέλουμε να εντάξουμε το μηχανισμό στο ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο, αλλά μέχρι τότε ε, υποστηρίζουμε μία πιο περιορισμένη μεταρρύθμιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας εν ώψη και του Συμβουλίου του Δεκεμβρίου και ε, των αποφάσεων που θα ληφθούν εκεί. να επισημάνω ότι κάποια από τα προβλήματα που αναφέρονται εδώ μάλλον δεν υφίστανται αυτή τη στιγμή. Υπήρξαν παρατηρήσεις για τον ε, διακυβερνητικό χαρακτήρα ε, του μηχανισμού σταθερότητας. Αυτό δεν θα αλλάξει στο εγγύς μέλλον. το πρώτο βήμα της ε, μεταρρύθμισης θα διατηρήσει τον διασυνοριακό διακυβερνητικό χαρακτήρα. Οπότε ήδη απολύονται τα ζητήματα των συνταγματικών περιορισμών και το καθεξής. Μπορεί να υπάρχουν ζητήματα σε περίπτωση ένταξης του μηχανισμού στο ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο. Το ίδιο ισχύει και για το θέμα της αιρεσιμότητας και στήριξης προς τα κράτη-μέλη. Σύμφωνα με το σχέδιο έκθεσής μας, είναι σαφές ότι ε, η πρωταρχική το πρωταρχικό μέλημα του μελλοντικού μηχανισμού θα πρέπει να είναι η παροχή συνδρομής στα κράτη-μέλη, αλλά βάσει του συμπεφωνημένου προγράμματος. Διατηρείται λοιπόν αυτή η ρητή αναφορά και στην έκθεσή μας. Ήθελα να πω ότι το πιο σημαντικό για το εγγύς μέλλον, τι πρέπει να περιμένουμε δηλαδή, είναι αφενός η δημιουργία του μηχανισμού ασφαλείας, του backstop, ως ένα ε, ενιαίο ταμείο εξυγίανσης που θα συμβάλλει στην ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης και στη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας και του Μελλοντικού Ταμείου Σταθερότητας και τη σχέση μεταξύ αυτού του θεσμικού οργάνου και του Κοινοβουλίου μας. Πρέπει να υπάρχει πολύ καλή συνεργασία μεταξύ των δύο οργάνων. Θα είναι ένα βήμα ε, προς ε, την αύξηση της ε, λογοδοσίας και δημοκρατικής νομιμοποίησης που συνάδουν και με τις περαιτέρω βελτιώσεις για την συνεργασία στον τομέα της οικονομικής διακυβέρνησης της Ευρωζώνης. Ο κύριος Μάνκα. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για τις παρεμβάσεις τους, για τα θετικά τους ε, σχόλια. Υπήρξαν και ορισμένες επικρίσεις και θα ήθελα να σταθώ εν συντομία σε αυτές. Είπατε ότι το ευρώ ε, δεν ε, αποτελεί επιτυχία μέχρι τώρα. Να σας υπερθυμίσω ότι χάρη στον μηχανισμό σταθερότητας, το ευρώ είναι πολύ πιο ανθεκτικό από οποιαδήποτε στιγμή στο παρελθόν. Επίσης, η στήριξη των πολιτών προς ε, το ευρώ ε, βρίσκεται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα από το 2002 και μετά. Σε σχέση μάλλον με την προηγούμενη περίοδο από το 2002 και μετά. Ε, βλέπουμε λοιπόν ότι οι προσπάθειές μας αποδίδουν. Αυτά για να απαντήσω στις επικρίσεις προς το ευρώ. Και κάτι άλλο. λέτε ότι εμείς θα ρίξουμε χρήματα σε ένα ταμείο, αλλά όχι. Θα αξιοποιήσουμε χρήματα που ήδη υπάρχουν και ο ίδιος ο μηχανισμός σε συνεργασία με την Επιτροπή θα κρίνει κατά πόσο πρέπει κάτι να αυξηθεί ή όχι. Αλλά όλα αυτά ε, υπόκεινται στην αυτοτέλεια αυτού του νέου θεσμικού οργάνου. Και σε αυτή την περίπτωση σίγουρα θα υπάρξει διαβούλευση και με το Κοινοβούλιο. Επόμενο σημείο. Σύμφωνα με τη συνθήκη, το νέο ταμείο δεν πρέπει να επαναλαμβάνει δραστηριότητε αρμο... Ε, αποκλειστική αρμοδιότητα των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων σε ό,τι αφορά την ε, εποπτεία των οικονομικών πολιτικών. Αυτέ ε, οι αρμοδιότητε παραμένουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Από νομική άποψη, είναι πολύ σημαντικό η Κομισιόν να διασφαλίσει ότι η ευρύτερη αξιολόγηση τη οικονομική κατάσταση στα κράτη-μέλη να συνάδει με τους κανόνες του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και για αυτό που είπατε για την ανάγκη προληπτικών μέτρων. Είναι κέρια σημασία αυτό το στοιχείο. Πρέπει να έχουμε προληπτικά μέσα και προληπτικές γραμμές, αν θέλετε, για εκείνα τα ε, κράτη-μέλη που έχουν καλύτερη δημοσιονομική εικόνα, ακολουθούν το σύμφωνο σταθερότητας ε, και ανάπτυξης έχουν πρόσβαση στις αγορές, δεν έχουν ζήτημα αφαιρεγγιότητας τραπεζών, όμως χρειάζεται πιστοτική γραμμή και για εκείνε τι χώρες που δεν ακολουθούν κάποια από τα κριτήρια ε, επιλεξιμότητας κάποιες χώρες μπορεί να πάρουν τέτοιες ε, γραμμές, όπως η Πορτογαλία, η Ελλάδα, η Ισπανία, η Κύπρος. Αλλά αυτές οι χώρες θα είναι υποχρεωμένες να υιοθετήσουν μέτρα για την βελτίωση της κατάστασης, ούτω ώστε να μετριαστούν οι κίνδυνοι ε, και να αποφύγουμε και τυχόν επιπρόσθετους ε, δυσκολίες χρηματοδότησης. Ευχαριστώ και θα παραδώσω τώρα την Προεδρία ξανά στον αγαπητό συμπρόεδρο. Ευχαριστώ, δεν έχω και πολλά να πω. Προθεσμία για τροπολογίες 9 Ιανουαρίου. 29 Ιανουαρίου θα εξεταστούν οι τροπολογίες. Οι επιτροπές μας θα ψηφίσουν 29 Ιανουαρίου, Ολομέλεια τον Φεβρουάριο. Η συνεδρίασή μας ε, συνεχίζεται αύριο στις 11. Λύεται αυτή η συνεδρίαση και θα συνεχίσουμε με την συνεδρίαση Econ Tax 3. Σας ευχαριστώ που ήρθατε.